Συνάδελφοι, χαίρετε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Θα κρατήσουν πολύ όπως ξέρετε και αφορούν ε, θεσμικά ζητήματα του Κοινοβουλίου, τον προπολογισμό. Ξεκινάμε λοιπόν ε, με το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017. Ζήτησαν το λόγο οι δύο εισηγητές για τον προπολογισμό της Ένωσης, του Κοινοβουλίου συγκεκριμένα, να ακούσουμε ευθύ αμέσω τον κύριο Γκάγερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητάω για